Chers collègues, je vous propose de, de prendre euh, place. Η Πρόεδρος. <clears throat> Καθίστε παρακαλώ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ευχαριστώ τον κύριο Γιούνκερ που πιστός στις ανταλλαγές απόψεών μας είναι πάλι σήμερα εδώ κοντά μας. Παρακαλώ τους Λουξεμβουργίους να καθίσουν. Όπως μου λέει ο πρόεδρος του Eurogroup. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Eurogroup, κύριο Γιούνκερ, που ήρθε σήμερα εδώ. Προφανώ η τελευταία ανταλλαγή απόψεων μα κατά τη διάρκεια τη ιδέα αυτή θα είναι. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε έναν τακτικό πλέον ρυθμό συζητήσεων δύο φορές το έτος για πολλά σημαντικά θέματα. Πολλά σημαντικά έγιναν με την τελευταία ανταλλαγή απόψεων που είχαμε προβήκατε σε μια σειρά δηλώσεων που συνέβαλαν στην κινητοποίηση των δημόσιων συζητήσεων και στις δικές μας εργασίες. Ε, υπάρχουν θέματα επί των οποίων συμπνέουμε και σίγουρα υπάρχουν θέματα που θέλουμε, μας ενδιαφέρει να έχουμε την αξιολόγησή σας. Η προετοιμασία του G20 και η σημασία που μπορεί να έχει την Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς είναι καθοριστικά, αλλά και οι συζητήσεις που ανακύπτουν για τις διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ χωρών μελών εντός και εκτός της ζώνης ευρώ, της αλληλεγγύης μεταξύ των δύο ενωτήτων και με το υποφόσκον ζήτημα που περάσαμε στα κείμενά μας ιδιαίτερα στην έκθεση που είχα συντάξει μας με τον κύριο Λάγκεν και που επανελήφθηκε σε πιο πρόσφατη ψηφοφορία και που αναφερόταν στο θέμα των Eurobonds, των ευρωομολόγων. Ένα θέμα επί του οποίου, ενός θέματος επί του οποίου λάβατε θέση και στο οποίο θα μπορούσατε να συμπληρώσετε τις απόψεις σας σήμερα. Ξέρετε το θέμα, προφανώς οι ερωτήσεις θα επαναφέρουν και άλλα ζητήματα συζήτηση. δίνω το λόγο και μετά θα έχουμε την συνηθισμένη ανταλλαγή απόψεων. Κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, όταν σας άκουσα να μου λέτε ότι είναι η τελευταία φορά που θα εμφανιστώ, που θα μιλούσα ενώπιον σας, φοβήθηκα κάπως, γιατί έχουμε εκλογές σε 7 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο. Εθνικές εκλογές. Και φοβήθηκα ότι δεν θέλετε να με ξαναδείτε μετά. Ελπίζω να επανεκλεγώ και να επανέλθω και ελπίζω επίσης, μια και έχουμε ευρωεκλογές την ίδια μέρα, να σας ξαναδώ όλους ή τους περισσότερους από εσάς, εσάς κυρία Πρόεδρε, ιδίως, που θέλω να ευχαριστήσω για την φιλοξενία που μου προσφέρατε τα τελευταία 4-5 χρόνια. Μετά την τελευταία μας συνάντηση στις 4 Νοεμβρίου του 8, όπως και εσείς είπατε, πολλά πράγματα έγιναν. Τα νέα διαφέρουν όλο ένα και περισσότερο. Επιδεινώνεται η οικονομική τα, τα νέα γίνονται χειρότερα και η οικονομική κατάσταση στην Ευρωζώνη όλο ένα και ταχύτερα επιδεινώνεται και αυτή, ενώ οι οικονομικές αγορές παραμένουν τότε Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν όλα τα κράτη της Ευρωζώνης, συμφώνησε τον Δεκέμβριο του 8 στη δημιουργία ενός κουτιού με μιας εργαλειοθήκης, ενός ε, συνόλου μέσων και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη για να καταπολεμήσουν σε ευρωπαϊκό πλαίσιο την ύφεση συμπληρώνοντας τα ευρωπαϊκά μέτρα με τα ενδεδειγμένα εθνικά μέτρα. Στο πλαίσιο αυτού του οικονομικού συστήματος ανάκαμψης της οικονομίας, τα κράτη-μέλη της Ένωσης ξεκίνησε να ε, υιοθετεί μέτρα σταθεροποίησης 3,5% του ΑΕΠ σε μέγιστο επίπεδο με έναν μηχανισμό αυτόματου σταθεροποιητή έχουμε και, άλλες, και άλλα μέτρα στη διάθεσή μας υψηλότερο επίπεδο. Μην περιμένετε το πρόγραμμα αυτό να δώσει άμεσες συνέπειες. Οι συνέπειες θα γίνουν αισθητέ σε βαθμιαίο τρόπο και ο αντίκτυπος των εθνικών μέτρων των προγραμμάτων ανάκαμψης θα γίνουν αισθητά κυρίως το 2010 και λιγότερο βραχυπρόθεσμα. Η οι οικονομικέ προβλέψεις, όπως έλεγα στο ξεκίνημα, συνεχίζουν να είναι πολύ κακές και συνεχίζουν να αναθεωρούνται προς τα κάτω. Η ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπή ε, της 7 Ιανουαρίου προέβλεπε μείωση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 1,9% το 2009 και μία μικρή ανάκαμψη 0,4% το 2010. Λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης. Ωστόσο, οι οικονομικές προβλέψεις αναφερούνται ακόμη περισσότερο προς τα κάτω. Οι τελευταίες εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ε, λένε ότι το ΑΕΠ της ζώνης ευρώ θα μειωθεί κατά 3,2% το 2009 και η, ανα, άνοδος το 2010 θα ήταν μόνο 0,1%. Στα πλαίσια της αποστολής του άρθρου 4 του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου του Όρθου 4 ήρθαν, ε, επισκέφτηκαν εκπρόσωποι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο Λουξεμβούργο και μου είπαν ότι οι αρμόδιες δομές του δούνου του αναθεωρούν ακόμη περισσότερο προς τα κάτω τα στοιχεία που είχαν αναγγείλει πριν από λίγους μήνες. Η κατάσταση της αγοράς εργασίας αντικατοπτρίζει αυτή την κακή οικονομική κατάσταση η ανεργία στο σύνολο της ζώνης ανέρχεται στο 8,2%. 13 εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς δουλειά. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η κατάσταση της αγοράς εργασίας που είχε βελτιωθεί σημαντικά κατά τα 10 πρώτα έτη ύπαρξης του ευρώ σκοτεινιάζει όλο και περισσότερο. Η κρίση της απασχόλησης, δεν μπορούμε να την πούμε και με διαφορετικό τρόπο, είναι προφανώς δραματική από πολλές οπτικές γωνίες και ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει με τον κάθε άνεργο ατομικά. Είναι προφανές ότι η κρίση της απασχόλησης θα οδηγήσει σε αντίξωες συνέπειες και σε επίπεδο δημόσιων οικονομικών, γιατί χρησιμοποιούμε τους αυτόματους σταθεροποιητές. Έτσι αποφασίσαμε. Επίσης, η αύξηση της ενεργείας σίγουρα θα έχει επιπτώσεις διαφορετικού και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα. Θα έχει μεταξύ άλλων συνέπειες και στην πιθανή ανάπτυξη η οποία θα μειωθεί. Επιπλέον, η, αύξηση, ισχυρή αύξηση της ενεργείας θα έχει αρνητικές συνέπειες και σε θέματα κοινωνικής συνοχής, στην ρήξη του κοινωνικού ιστού και αυτό θα οδηγήσει προφανώς σε πολιτικούς, σοβαρούς και προφανείς πολιτικούς κινδύνους. Στο Eurogroup το Φεβρουάριο είχαμε μια πρώτη συζήτηση για την κατάσταση στην αγορά εργασία στο χώρο ευρώ. Οι Υπουργοί Οικονομικών της Ζώνης Ευρώ ενδιαφέρονται από κοντά για τις συνέπειες της κρίσης στην απασχόληση και συμπεράναμε ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που υιοθετήθηκαν μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής της Λισαβόνας είναι απαραίτητες, όμως αυτές οι μεταρρυθμίσεις που έχουν στόχο ε, μέσο πρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ε, πρέπει να συμπληρωθούν και με βραχυπρόθεσμες προσπάθειες που θα έχουν σαν στόχο να διατηρήσουν αν θέλετε κάπως την ε, οικονομία και να ε, ενθαρρύνουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία να χρησιμοποιεί περισσότερο την μερική απασχόληση αν θέλετε και όχι τις ε, απολύσεις. Και εξετάσαμε και τις διαφορετικές μορφές ε, της μερικής ανεργίας, την, τα επιδόματα ανεργίας που θα πρέπει να συμπληρωθούν με, ένα, με μια πιο αυξημένη, με ένα πιο αυξημένο επίπεδο των εργαζομένων που συμμετέχουν σε ε, προσπάθειες κατάρτισης, συμπληρωματικής κατάρτισης, ενώ βρίσκονται σε τεχνητή ανεργία. Οι κυβερνήσεις τώρα αποφάσισαν να βοηθήσουν, αν θέλετε, να προσφέρουν, να συνεισφέρουν στο κεφάλαιο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με ε, ένα σημαντικό ποσό και έχουμε ε, επίσης ε, αποφασίσει ένα νομοθετικό πλαίσιο για αυτά τα, τοξικά προϊόντα τα οποία έχουν πληθύνει παρά τις προσπάθειες, παρά την πλαισίωση κτλ. Η, η εμπιστοσύνη επιστρέφει πάρα πολύ αργά και ε, υπάρχει μία έλλειψη εμπιστοσύνης στην πρόσβαση, στην πίστοση αν θέλετε. Ακόμα δεν έχει βρεθεί μία απάντηση ικανοποιητική γιατί κάθε πιθανή λύση έχει σημαντικές ε, συνέπειες ε, στις, στην, στα δημόσια οικονομικά και ε, θέτει σημαντικά προβλήματα στα θέματα ισότητας και ε, ισότιμης συνεισφοράς όλων των φορολογουμένων. Και όλα αυτά τα τοξικά προϊόντα ε, κινδυνεύουν να δημιουργήσουν ηθικά αν θέλετε προβλήματα αλλά και πιθανές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και σε όλα αυτά τα προβλήματα δεν υπάρχει μία ενιαία απάντηση. Παρ' όλα αυτά όμως πιστεύουμε, λένε και περισσότερο, ότι αν δεν υπάρχει μια κατάλληλη μεταχείριση των τοξικών προϊόντων θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επανέλθει η εμπιστοσύνη στην χρηματοπιστωτική αγορά και η επιστροφή της εμπιστοσύνης ε, είναι απαραίτητη έτσι ώστε να ε, αρχίσουν να ρέουν πάλι οι πιστώσεις. Όλες αυτές οι εξελίξεις, ε, τις οποίες ε, σας ανέφερα αλλά και άλλες ακόμα, θα οδηγήσουν σε, μεσοπρό... σε βράχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και ε, μακροπρόθεσμους συνέπειες στο δημόσια έλλειμμα, δημόσιο έλλειμμα η Κομισιόν πιστεύει ότι το έλλειμμα από 1,7 το 2008 θα φτάσει στο 4.000 το 2009 και θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο το 2010. Το δημόσιο χρέος των κρατών μελών μέχρι το 2010 η Κομισιόν πιστεύει ότι θα φτάσει στο 76% του ΑΕΠ της ε, ζώνης ευρώ. Το δημόσιο χρέος. Η... Το έλλειμμα μπορεί να... Οι προβλέψεις λένε ότι θα μειωθεί, αλλά τα... το χρέος θα αυξηθεί. Η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρεί στην ενδιάμεση αξιολόγηση ότι από τα νέα κράτη, τα νέα κράτη-μέλη από τα 16 της ζώνης ευρώ θα έχουν ένα δημόσιο έλλειμμα ε, το οποίο θα ξεπερνάει το 3% το 2009. η κατάσταση δεν βελτιώνεται γιατί οι προβλέψεις ε, σκοτεινιάζουν αν θέλετε, γίνονται όλα ένα και πιο δυσμενείς και το Eurogroup στην συνεδρίαση της αρχές Μαρτίου θεωρούσε ότι θα ήταν, ε, δεν θα ήταν σκόπιμο να ε, υιοθετήσει συμπληρωματικά μέτρα. Πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανακαμψής δεν απαιτεί συμπληρωματικά μέτρα και αυτή η άποψη εκφράστηκε από, την, ε, από το Eurogroup και επιβεβαιώθηκε και από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στο Εαρινό Συμβούλιο, στην Εαρινή Σύνοδο Κορυφής. Ε, είπαμε ότι θα πρέπει, δεν θα πρέπει να υιοθετηθούν συμπληρωματικά μέτρα, διότι, γιατί τώρα θα πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι συνέπειες των μέτρων που έχουμε ήδη υιοθετήσει. Επίσης, ανησυχούμε όλο ένα και περισσότερο για τις συνέπειες αυτού του προγράμματος ανάκαμψης στα δημόσια, στην δημόσια οικονομία και αν το έλλειμμα διευρυνθεί ή το, αυτό, το χρέος αυξηθεί, θα πρέπει... Θα δούμε ότι οι πολίτες θα χάσουν την εμπιστοσύνη τους, διότι τα, τα ελλείμματα τώρα είναι οι φόροι του αύριο. Επομένως ε, πρέπει να, είμαστε, να επαγρυπνούμε πάνω στο σημείο αυτό, κυρίως διότι δεν αγνοούμε και τις συνέπειες του crowding out που έχει να κάνει το μεγάλο δημόσιο χρέος και κάποιες επιχειρήσεις ε, ήδη το συναισθάνονται αυτό. Τώρα, το Σύμφωνο Σταθερότητας ε, και Ανάπτυξης που που μεταρρυθμίστηκε το 2005, ανέχεται κάποια δημόσια ελλείμματα τα οποία ξεπερνούν το 3% εφόσον αυτή η υπέρβαση του 3% είναι προσωρινή, εστιασμένη και κοντά αν θέλετε στην αξία αναφορά, στην τιμή αναφοράς. Ε, συνειδητοποιούμε επομένως το γεγονός ότι βράχει πρόθεσμα, δεν έχουμε άλλες αναλλακτικέ λύσεις παρά μόνο να διευρυνθεί το έλλειμμα όμως συνειδητοποιούμε ότι βράχει πρόθεσμα, ακολουθούμε μία πολιτική η οποία είναι καλή μεν, αλλά είναι κακή στο, σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Επομένως θα πρέπει άμεσα όσο το πιο γρήγορα να υιοθετήσουμε μια στρατηγική εξόδου από αυτή την κατάσταση που θα μας επιτρέψει να ε, καταλήξουμε σε μια δημοσιονομική εξυγίανση. Τώρα, η έναρξη των διαδικασιών ε, που αφορά την υπέρβαση του δημοσίου ελλείμματος, δηλαδή στη Γαλλία, στην Ισπανία και στην, στην Ελλάδα και στην, Πορτογα... Ιρλανδία, ε, θα συζητηθούν στην Πράγα, στη Σύνοδο Κορυφής της Πράγας και, το... και εκεί θα πρέπει να πούμε την άποψή μας για κάποια ενδεχόμενη στρατηγική εξόδου που θα πρέπει να υιοθετήσουμε. Το Eurogroup δεν συζήτησε την δυνατότητα να μην μπορέσει να εξασφαλίσει τις πληρωμές ένα κράτος μέλος της ζώνης ευρώ. Βέβαια κάτι τέτοιο αναφέρεται συχνά και στις, στο δημόσιο τύπο και στις συζητήσεις μας, διότι ε, θεωρούμε ότι ο κίνδυνος ε, ένα κράτος μέλος να εγκαταλείψει τη ζώνη ευρώ και να επανεισάγει το εθνικό του νόμισμα θα μπορούσε να εξασφαλίσει έναν έλεγχο στα δικά του δημοσιονομικά δηλαδή, αυτό είναι κάτι, ένας, ένας ο οποίος δεν τίθεται. Τώρα, η πάυση πληρωμόνου, η στάση πληρωμόνου ενός κράτους μέλους της ζώνης ευρώ και αυτός δεν είναι ένας κίνδυνος τον οποίο αντιμετωπίζουμε θεωρούμε εμείς τουλάχιστον. Ε, κανένα κράτος μέλος της ζώνης ευρώ δεν αντιμετωπίζει μέχρι στιγμής δυσκολίες για να εξασφαλίσει μια χρηματοδότηση από την αγορά. Βέβαια, ορισμένα κράτη-μέλη έχουν ε, μεγάλο spread, εξασφαλίζουν χρηματοδότηση ε, δάνεια με μεγάλο spread σε σχέση με το Deutsche Mark. Βέβαια, υπάρχουν ε, θα πρέπει να υιοθετηθούν βραχυπρόθεσμα μέτρα, υπό τον όρο βέβαια δεν θα επηρεάσουν μακροπρόθεσμα την κατάσταση. Και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ούτως ή άλλως ε, έχει αναφερθεί σε διάφορα μέτρα και για, το, αυτή, την, για το είδος της ε, δανειοληψίας αν θέλετε με το spread που είναι ένα σύγχρονο μέτρο, ε, πολύ σύγχρονο. Υπάρχουν ε, κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες. Από την δημιουργία της ζώνης ευρώ είδαμε ότι Υπάρχουν διαφορές όσον αφορά τον ε, πληθωρισμό που άλλαξαν ε, την ε, κατάσταση στη ζώνη ευρώ και κάποια κράτη-μέλη έχουν αυξημένα ελλείμματα του τρέχοντος ισοζυγίου πληρωμών. Και αυτές οι διαφορές, οι αποστάσεις αν θέλετε, αντικατοπτρίζουν έναν κίνδυνο για την συνοχή της ζώνης ευρώ. Γι' αυτό τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν διαρθρωτικές πολιτικές που θα έχουν σαν στόχο να περιορίσουν ή να εξαφανίσουν αυτές τις διαφορές. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο η Ευρωζώνη αποφάσισε τον, ε, τον Ιανουάριο να κάνει ένα ε, τακτικό έλεγχο και παρακολούθηση τα, ε, όλων των θεμάτων που αφορούν την ανταγωνιστικότητα, διότι είναι θέματα τα οποία είχαμε υποτιμήσει το πρώτο, την πρώτη πενταετία της δεκαετίας του ευρώ. Τώρα, ένα ερώτημα το οποίο συζητάμε συνέχεια είναι η διεύρυνση της ζώνης ευρώ. Αυτό το ερώτημα, αυτό το θέμα συζητήθηκε πολύ όταν προσχώρησε η Σλοβακία στη ζώνη ευρώ και παρά τις, τα οικονομικά και δημοσιονομικά προβλήματα η Σλοβακία μπόρεσε να μπει στο ευρώ χωρίς κανένα πρόβλημα και θα πρέπει να συγχαρούμε τις σλοβακικές αρχές για, το, για την κατάσταση αυτή. Όμως θεωρούμε ότι θα ήταν επικίνδυνο αυτή τη στιγμή αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, όπως τα λέει ο κύριος Τρισέ, να ανοίξουμε ξανά τη συζήτηση για τα κριτήρια σύγκλησης. Ε, τα τελευταία χρόνια το κάνουμε αυτό πάρα πολύ συχνά και συζητάμε καταρχάς το αξιόπιστο του κριτηρίου του ελλείμματος, της, του χρέους, ε, της, ε, του πληθωρισμού και τώρα συζητά, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να ανασυζητήσουμε τώρα ξανά τα θέματα αυτά, ούτε για τα θέματα ισοτιμίας, ε, συναλλαγματικής ισοτιμίας. Αυτό το οποίο έκανε όμως ε, το Eurogroup το Μάρτιο ήταν να μην ανοίξει ξανά η συζήτηση αυτή, διότι θεωρούμε ότι η σταθερότητα της ζώνης ευρώ δεν είναι ένα δημιούργημα το οποίο έπεσε έτσι από τον ουρανό, δεν, είναι, δημιουργήθηκε εκ του μηδενός ή αυθορμήτως, αλλά είμαστε ε, πεπισμένοι ότι η σταθερότητα των οικονομικών ε, αποτελεσμάτων είναι συνετή και πρέπει να προσανατολίζεται σε μια σταθερότητα τα θέματα σύγκλησης ε, και η σταθερότητα των κριτηρίων σύγκλησης, αν θέλετε, ε, συνεισφέρουν σημαντικά στην γενικότερη σταθερότητα. Το Ευρωγκρούπ και η Ευρωζώνη δεν ε, είναι ένα κλειστό όμιλο. Το γεγονος οτι ότι τέσσερα κράτη-μέλη προσχώρησαν στην Ευρωζώνη προφανώς αποδεικνύει ότι όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης που πληρούν τα κριτήρια μπορούν να έχουν και οφείλουν να έχουν προσχώρηση ή είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιήσουν το δικαίωμα προσχώρησης τους στην ζώνη ευρώ. Και θα ήθελα να εδώ να επωφεληθώ για να πω δύο λόγια για τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ο τρόπος παρουσίασης των πραγμάτων που διαιρεί την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ομάδες δεν με βρίσκει σύμφωνο. Δηλαδή τον χωρισμό της Ευρώπης στη Δυτική Ευρώπη δηλαδή ενάρετα μέλη και την Ανατολική Ευρώπη κακά μέλη. Πρόκειται για μια περιγραφή που θυμίζει την σοβιετική διαίρεση της ε, υπήρου της Ευρώπης. Δεν υπάρχουν μπλοκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κράτη-μέλη που έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις, τα ίδια. Και άλλωστε το κεντρικό και ανατολικό τμήμα της Ευρώπης όπως έχετε διαπιστώσει περιλαμβάνει τελείω διστάμενε καταστάσεις μεταξύ των κρατών μελών. Δεν μπορεί να υπάρξει μια έτοιμη στρατηγική για όλες τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, αλλά να λαμβάνουμε υπόψη τις, τα ειδικά χαρακτηριστικά των μεν και των δε. Με ρωτήσετε πρόεδρε για την προετοιμασία του G20. Κάναμε κάποιες ανταλλαγές απόψεων στο Eurogroup, ακόμα περισσότερο στο ECOFIN, ακόμα δε περισσότερο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Άλλωστε το Eurogroup δεν είναι μέλος το, του G20, αλλά που δεν είναι πια ούτε καν G20, G22, G23, είναι μνήκη κομισιόν μέσα. Εγώ Έχω την εντύπωση πάντως ότι το G20 είναι μια πιο αντιπροσωπευτική και δημογραφικά ισορροπημένη δομή από ότι το G7 ή το G8, αλλά διαπιστώνω ότι τα κράτη που δεν μετέχουν στο G20 δυσκολεύονται να ενημερώνονται παρκώς όσο τουλάχιστον και οι μετέχοντες στο G20. Είχα συναντήσει την κυρία Μέρκελ στην προπαρασκευαστική συνάντηση των κρατών της Ένωσης που είναι μέλη στο G20, καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα που πέρασαν στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου. Από πλευράς μου θέλω να τονίσω ότι δεν θα ήθελα να, τέξει, να τέκει μην η ε, η συνάντηση του G20 και δεν θα ήθελα να γίνει η ομάδα αυτή ε, μια δομή που θα χωρίσει αυτούς που κάνανε πάρα πολλά και αυτούς που δεν έχουν κάνει αρκετά. Η συνάντηση θα πρέπει να έχει σαν κύριο στόχο τη διαμόρφωση μιας νέας διεθνούς οικονομικής αρχιτεκτονικής. Αυτά ήθελα να σας πω Τώρα φαντάζομαι ότι οι συνάδελφοι ε, θα θέσουν άλλα ερωτήματα στα οποία θα απαντήσω όσο περισσότερα μπορώ. Ευχαριστώ. Έχω ένα μεγάλο κατάλογο μιλητών. Αυξάνει το κατάλογος. Προτείνω να είσαστε λυτοί στις παρεμβάσεις. Η κυρία Ελίζα Φερέρα και μετά ο κύριος Βολφ Κίτς. Thank Σας ευχαριστώ. Θα τα πω στα αγγλικά. Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ κύριε Πρωθυπουργέ. Ήθελα να υπενθυμίσω ότι κάθε μέρα οι προβλέψεις είναι και χειρότερες. Το, ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος που δημοσιεύθηκε μόλις πρόσφατα προβλέπει τα χείριστα σχετικά με το κλίμα του επιχειρήν. Και ο ΩΣΑ στην πιο πρόσφατη διάσκεψή του διορθώνει προς τα κάτω πάλι <clears throat> τις προβλέψεις για την ε, ανάπτυξη στην Ευρώπη και μάλιστα μείον 3% ακόμα χειρότερα και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Παρ' όλα αυτά, εσείς αναφέρατε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι οι αποκλήσεις μεταξύ χωρών και ότι η ικανότητα κάθε χώρας να αντιδράσει στις εξελίξεις αυτές είναι από τις πιο ε, μεγάλες και ότι αυτό είναι απόρρια του κοινού νομίσματος και επίσης είπατε ότι δεν υπάρχει λόγος να επανατεθεί επιτάπητος το σχέδιο ανοικοδόμησης. Βέβαια γνωρίζετε ότι αυτό το σχέδιο συναποτελείται από τα εθνικά σχέδια ανάπτυξης ή αποκατάστασης. Και μάλιστα ακυρώσατε και την διάσκεψη κορυφής για την απασχόληση. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει ε, κάποιο οριζόντιος μηχανισμός, ακόμα και εκείνες τις ε, χώρες, οι οποίες δεν έχουν κανένα εργαλείο στην εργαλειοθήκη τους. Ε, δεν προβλέπεται καμία οριζόντια πρωτοβουλία για να αντιμετωπιστούν τα πράγματα. Και τι γίνεται με τα ευρωομόλογα. <clears throat> Τέλος, για το G20. Το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσε να γίνει θα ήταν να μην γίνει απολύτω τίποτα στο G20. Αφενός δηλαδή ο αγώνας κατά των φορολογικών παραδείσων και τα λέω ομά λίγο, αλλά νομίζετε ότι η ευρωπαϊκή θέση στο G20 δεν θα τεθεί σε κίνδυνο αφού ακόμα έχουμε μέσα στην ίδια την Ευρώπη φορολογικούς παραδείσους και απόρριτο τραπεζικών λογαριασμών και μόλις ψηφίσαμε εμείς την κατάργηση του απορρίτου μέχρι το 2014 δηλαδή μετά από μακρό και δύσκολο αγώνα. Ποιες είναι οι θέσεις σας για τα θέματα αυτά. Βολφ Κλίντς και μετά Γκάι Μίτσελ. Κύριε Πρόεδρε, όλοι γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζουμε σοβαρή κρίση εμπιστοσύνης. Η παγκόσμια οικονομία έχει παραλύσει και όλοι οι παρατηρητές θεωρούν ότι για να επανέλθουμε σε ομαλή κατάσταση, να αρχίσουν δηλαδή να λειτουργούν και πάλι οι τράπεζες κτλ. Αυτό θα περάσει καιρός. Μία πάντως από τις προϋποθέσεις είναι ότι πρέπει να επιληθεί το θέμα των τοξικών προϊόντων. Ο Γκάιτνερ την προηγούμενη εβδομάδα παρουσίασε το σχέδιό του, δηλαδή πώς ε, σχεδιάζει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στι Πολιτείε. Μπορεί να μην είναι το σοφότερο πράγμα που έχουμε ακούσει ποτέ, αλλά είναι μια πάντω προσπάθεια να κάνει κανεί κάτι. Εσεί είπατε ήδη ότι στην Ευρώπη δεν έχουμε ακόμα συγκεκριμένη προσέγγιση ούτε επιμέρου αλλά ούτε στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ερωτήσει. Πρώτον, ω πρόεδρο τη Ευρωομάδα, δεν θεωρείτε ότι είναι κατά, κατεξοχήν καθήκον σα στους καιρούς αυτούς να φροντίσετε ώστε να υπάρξει μια προσέγγιση εναρμονισμένη στο ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Και επειδή δεν το έχουμε αυτό το πράγμα, δεν φοβάστε ότι στο G20 θα αντιμετωπίσετε ε, βαριά και μαζική κριτική από τους υπολείπους. Δεύτερον, είπατε ότι 9 από 16 χώρες της ευρωομάδας, της ε, ζώνης ευρώ, είναι σαφώς άνω του 3% και δεν πληρούν και τα άλλα κριτήρια. Πώς θα επανέλθουμε σε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς εφόσον αντιμετωπίζουμε τους αμαρτωλούς, ας πω έτσι, όπως και στο παρελθόν. Γιατί στο παρελθόν υπήρξαμε πολύ γενναιόδοροι απέναντι στους αμαρτωλούς. Για παράδειγμα, δεν καταδικάσαμε τη Γερμανία, παρόλο που για πολλά χρόνια παραβίαζε το σύμφωνο. Μήπως πρέπει να επιβάλλουμε πολύ συγκεκριμένες κυρώσεις, ώστε να συμμορφωθούν όλοι αυτοί. Τελευταίο, δεν φοβάστε ότι με αυτά τα τεράστια κενά, τα τεράστια δημοσιονομικά κενά, σε λίγα χρόνια θα αντιμετωπίσουμε καλπάζοντα πληθωρισμό. Και πώς νομίζετε ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε το ενδεχόμενο αυτό. Ευχαριστώ. Τελευταίος αυτών των πρώτων τριών, Γκάι Μίτσελ. Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται ψυχραιμία και προσεκτική προσέγγιση. Ούτε θέλω να δω μια λύση η οποία να επιδεινώσει τα πράγματα. Νομίζω ότι βρισκόμαστε στην κατάσταση αυτή επειδή χάσαμε λίγο τους στόχους μας από τα μάτια μας. Στην πραγματικότητα πρώτα έπρεπε να εκενώσουμε τα τέλματα και να ρίξουμε περισσότερο βάρος στην ανάκαμψη Ναι, μεν πρέπει να σβήσουμε τη φωτιά τώρα, αλλά πρέπει να φτιάξουμε και τον πυροσβεστικό σταθμό για το μέλλον. Ετοιμαζόμαστε για την ανάκαμψη. Είναι ευκαιρία τούτο εδώ, η παρούσα κρίση, για να γίνουμε και πιο ανταγωνιστικοί. Άκουσα ότι το σχέδιο ανάκαμψη δεν χρειάζεται ειδικά μέτρα. Ενώ, εννοεί φαντάζομαι ότι δεν χρειάζονται πρόσθετα μέτρα από πλευρά χωρών μελών. Αλλά δεν υπάρχει Χώρο για να λάβει πρόσθετα μέτρα, για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και θα μπορούσε ο πρόεδρος Γιούνκερ να μας πει τι συζητήσει διεξάγονται με την Κίνα. Εγώ πέρασα από την Κίνα πρόσφατα και έγινε εκεί υψηλού επίπεδου διάσκεψη ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας στο Πεκίνο λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Ποιες ευκαιρίες υπάρχουν συνεργασίας μεταξύ Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωση για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Εγώ νομίζω ότι επαφιέμεθα υπερβολικά στις επιμέρους προσεγγίσεις των χωρών μελών. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να εμπλακεί και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά και να ε, τονωθούν οι σχέσεις με, την, με άλλες χώρες όπως η Κίνα για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί καλύτερα η κρίση. Κυρίε και κύριοι, έχετε την εντύπωση ότι θέσατε τρεις ερωτήσεις, αλλά θέσατε δέκα ερωτήσεις τουλάχιστον. Η, κυρίως, η κυρία Φερέιρα Είσαστε ανεξάντλητοι, διότι σε δύο λεπτά έθεσε πέντε ερωτήσεις. Και εγώ σε δύο λεπτά θα απαντήσω και στις δέκα ερωτήσεις. Θα επιλέξω βέβαια αυτές τις ερωτήσεις που με βολεύουν. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι πιστεύω ειλικρινά ότι δεν χρειαζόμαστε, δεν χρειάζεται να αυξήσουμε τον όγκο, αν θέλετε, του προγράμματος ανάκαμψης. Το ευρωπαϊκό κομμάτι είναι πολύ στενό, αν θέλετε. Περάσαμε 4-5 μήνες για να συζητάμε αν για το κατά πόσο θα πρέπει να ε, ε, χρησιμοποιήσουμε 5 δισεκατομμύρια ευρώ και αν τα χρησιμοποιήσουμε ε, σε τι χρήση θα τα, θα χρησιμοποιήσουμε, που θα τα πάρουμε και όλα αυτά, νομίζω ότι γίναμε γελοί. Και πιστεύω ότι το ευρωπαϊκό κομμάτι, αν θέλετε, μπορεί να, πρέπει να είναι σημαντικό, αλλά τα κράτη-μέλη και έχουν υιοθετήσει εξαιρετικά μέτρα όσον αφορά τουλάχιστον την φιλοδοξία των μέτρων και την, το μέγεθος των μέτρων. Τώρα, εάν προσθέσετε όλα όσα συμμετέχουν, θα φτάσει στο 23% του ΑΕΠ. 23% του ΑΕΠ. Εάν προσθέσετε δηλαδή στους αριθμούς αυτούς και τα, τα ποσά για τις εγγύσεις και τα λοιπά, αλλά θα δείτε ότι φτάνουμε στο 23%. Τα δημοσιονομικά μέτρα είναι 3 έως 4% του ε, ΑΕΠ και δεν απέχουν πολύ από τις προσπάθειες που ήδη έχουν υιοθετήσει οι Ηνωμένε Πολιτείε και πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να προσθέσουμε άλλα μέτρα εάν δεν αξιολογήσουμε, αν δεν μετρήσουμε τις συνέπειες των μέτρων που εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή τα Eurobonds τώρα. Αυτή είναι μια ιδέα που είχα ε, αναφέρει πριν από έξι μήνες. Θα τα συζητήσουμε και αυτά τα Ομόλογα και τώρα και στο μέλλον. Και κάποιοι συνάδελφοί μου δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι και ίσως φτάσει κάποια μέρα που Ίσως να μετανιώσουμε που δεν ακολουθήσαμε τη συνετή συμβουλή του Προέδρου της, του Eurogroup, διότι τα ευρωομόλογα μπορεί να μας ε, επέτρεπαν να αποφύγουμε κάποια ατυχήματα ή να διορθώσουμε την κατάσταση. Και τα ευρωομόλογα θα ε, είναι ε, χρήσιμα βέβαια ε, εφόσον υπάρχει βέβαια και μία ε, υπηρεσία αν θέλετε και ένας μηχανισμός σφαιρικής επίβλεψης. Εγώ είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό, σε αυτή την ιδέα. Τώρα, γιατί καταργήθηκε, ακυρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής για την απασχόληση. Να σας πω καταρχάς ότι δεν ακυρώθηκε. Απλώς ε, δόθη μια νέα διάσταση, αν θέλετε, στην, ε, στην, ε, στο μέγεθός της, αν θέλετε, διότι θα η Τρόικα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συζητήσουν τα θέματα απασχόλησης με τους κοινωνικούς εταίρους. Εγώ δεν είχα προτείνει την ιδέα να υπάρξει μια σύνοδος κορυφής ε, της, για την απασχόληση. Η μόνη σύνοδος κορυφής για την απασχόληση που έλαβε χώρα μέχρι τώρα ήταν μια σύνοδος κορυφής στην οποία, την οποία συμμετείχα και στην οποία προείδρευα ο κύριος Γκέμπελης ήταν παρόν και οφείλετε να ομολογήσατε ότι δεν ε, ε, εστέφθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία. Βέβαια, υιοθετήσαμε κάποιες κατευθυντήρες γραμμές για την απασχόληση. Το 1997 δεν λέω ότι αυτά τα οποία έκανα τότε ε, δεν ισχύουν ή κάναμε, ήταν ένα μηδενικό, αλλά το Συμβούλιο αποφάσισε να μην επανέλθει στα θέματα αυτά, είτε το Δεκέμβρη είτε το, την Άνοιξη. Είχαμε αποφασίσει από το 1997 ε, να υπάρχει ένα, μια σύνοδος κορυφής για την απασχόληση. Η, η Τσεχική Προεδρία είπε να έχουμε μια κοινωνική, μια κοινωνική σύνοδο κορυφής, διότι δεν έχει να κάνει μόνο με την απασχόληση, είναι και τα θέματα κοινωνική συνοχή ε, γενικότερα. Τώρα το Συμβούλιο, η Σύνοδο Κορυφή αποφάσισε να το ακυρώσει. Τώρα, ο Τσέχος Πρωθυπουργός δήλωσε ότι ότι οι πρωθυπουργοί που θέλουν να συμμετέχουν στην Τρόικα είναι ευπρόζεκτοι εγώ χαίρομαι για κάτι τέτοιο και θα ήθελα να πάρω μέρος, διότι νομίζω ότι το μήνυμα το οποίο είχαμε δώσει στην αρχή ε, ήταν θετικό. Τώρα όμως που, κάνουμε, που αλλάξαμε, αν θέλετε, την, την, τη σύνθεση αυτής της ε, συνάντησης, αν θέλετε, είναι ένα, ε, αυτό μήνυμα που στείλαμε είναι κακό για τους εργαζομένους και για τους άνεργους Τώρα, για τους φορολογικούς ε, παραδείσους, tax havens, το τραπεζικό απόρριτο. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν αφορά το Eurogroup. Έχω όμως κάποιες ιδέες πάνω στο θέμα. Διαπιστώσατε κι εσείς όπως και εγώ, αλλά εγώ το διαπίστωσα πριν από εσά, ότι οι διεθνείς τάσεις, τις οποίες παρατηρούμε εδώ και κάποια χρόνια, δείχνουν σαφέστατα ότι το τραπεζικό απόρριτο είναι ένας θεσμός, αν θέλετε, που χάνει τη σημασία του. Είδατε ότι η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κόνγκ και άλλοι έχουν εκδηλώσει το την, ε, την θέλησή τους να προχωρήσουν σε μια ανταλλαγή ε, πληροφοριών και το Βέλγιο και η Αυστρία και το Λουξεμβούργο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θέλουν να εφαρμοστεί η συνθήκη του ΟΣΑ, κυρίως όσον αφορά το άρθρο 26.5 που αφορά την ανταλλαγή των πληροφοριών. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο δεν τίθεται πλέον, διότι από εδώ και πέρα όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κάνουν αυτό που τους ζητάνε. Δηλαδή στις ε, συμφωνίες της διπλής φορολογίας θα αναφέρεται και το εργαλείο αυτό της ανταλλαγής των πληροφοριών κατόπιν αιτήματος. Δεν θα συνεχίσουμε τώρα να συζητάμε για ένα πρόβλημα το οποίο ούτως ή άλλως έχει βρει τη λύση του. Στη χώρα μου παραδείγματος χάρη ε, ασχοληθήκαμε με διάφορα απευθυνθήκαμε σε διάφορα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διεθνούς εταίρους έτσι ώστε να συμπληρώσουμε τις συμφωνίες διπλής φορολογίας στα θέματα και τα θέματα αυτά. Τώρα, μια και θα υπάρξει συζήτηση για τα θέματα συνεργασίας, όλα αυτά ε, θα πρέπει να θα πρέπει να το δούμε με ιδιαίτερη προσοχή το θέμα, διότι εγώ έχω την εντύπωση ότι δεν είναι ε, ένα-δύο τα τα ιδρύματα, αν θέλετε, και οι θεσμοί που ε, εμπλέκονται. Έχω μετρήσει 91 ε, θεσμούς ή υπηρεσίες ή οργανισμούς που εφαρμόζουν και θα ήθελα τα κράτη-μέλη τα οποία ε, κατηγορούν αν θέλετε τις, το Βέλγιο, την Αυστρία και, την, και το Λουξεμβούργο θα πρέπει να εφαρμόσουν την ίδια πρακτική και θα πρέπει να έχουν το θάρρος να εφαρμόσουν την ίδια πρακτική και με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Στις Ηνωμένε Πολιτείε, δεν υπάρχουν ξεχωριστές πολιτείες, υπάρχουν κάποια ε, κάποια νησιά αν θέλετε και αν ε, που δεν χρειάζεται να μάλλον να, μιλάμε για, για υπεράκτια ή για κάποια νησιά υπάρχουν και πολιτείες συγκεκριμένες και γι' αυτό, εάν υπάρξει κατάλογος, θα πρέπει να δούμε και τι θα γίνεται και με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Και πιστεύω, θα πρέπει να το θίξουμε το θέμα αυτό. Θα πρέπει ο κύριος Μπράουν να πει στον κύριο Ομπάμα να ε, βάλει ένα τέλος στους φορολογικούς παραδείσους που υπάρχουν στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. και θα δούμε μέχρι τι 3 Απριλίου, αλλά αυτά έγιναν για να εντυπωσιαστεί το κοινό ή για να δοθεί μια ουσιαστική λύση στο πρόβλημα, στο πραγματικό πρόβλημα που υπάρχει και στις Ηνωμένε Πολιτείε ακόμα. Τα τοξικά. Bad assets. Για τα τοξικά προϊόντα, τέλος πάντων, ε, δεν έχουμε μια έτοιμη λύση. Έχουμε προτείνει κάποιες, ε, κάποια εργαλεία, αν θέλετε, κάποιους περιορισμούς, κάποια caveats, αλλά πιστεύω ότι εάν δεν διορθωθεί η κατάσταση, δεν θα υπάρξει, αν δεν ε, υπάρξει μια ανόρθωση εμπιστοσύνης, επιστροφή της εμπιστοσύνης, δεν πρόκειται να υπάρξει ξανά ροή των πιστώσεων. Τώρα αυτό όμως είναι θέμα του ΕΚΟΦΗΝ. το ΕΚΟΦΗΝ θα πρέπει να δώσει μια απάντηση. Και μετά θα πρέπει να αξιολογήσουμε βέβαια λεπτομερώς τα υπέρ και τα κατά της αμερικανικής πρότασης. Διότι ακόμα είναι πάρα πολύ καινούρια για να την αξιολογήσουμε. Χρειάζεται να Ίσως ισοσκελιστούν οι προϋπολογισμοί. Μίλησα για μια στρατηγική εξόδου. Θα διατυπωθεί τους επόμενου μήνε. Πρέπει να δώσουμε την βεβαιότητα στους πολίτες ότι δεν πρόκειται να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και είμαι αντίθετος να αρχίσουμε πάλι να μιλούμε για κυρώσει γιατί σε αυτόν τον κύκλο της συγκυρία δεν έχει πολύ νόημα να επαπειλούμε κυρώσει ούτε έχει νόημα άλλωστε να προκαλέσουμε και άλλα προβλήματα ε, στην συγκυρία με ακόμα περισσότερους περιορισμούς στους προϋπολογισμούς. Αυτά δεν είναι άλλωστε πράγματα τα οποία πρόκειται να γίνουν σε ένα-δύο χρόνια. Θα εξαρτηθούν όμως και από την δημοσιονομική αφετηρία των χωρών εκείνων που ε, ξεπερνούν το 3%. Ο πληθωρισμός με ανησυχεί, όχι διότι υπάρχει τώρα, αλλά διότι είναι σημαντικός ο κίνδυνος στην, κατά την έξοδο από την κρίση. Δεν υπάρχουν όμως άλλα ιστορικά παραδείγματα, μπορεί να βρεθούμε ε, απέναντι σε έναν ισχυρό ε, πληθωρισμό. Ε, συνεχίζει τα γαλλικά πάλι. Την ναι. Κίνα στα, στον τελευταίο καιρό δεν είχαμε συγκεκριμένες ε, συναντήσεις ε, που να αφορούν ε, την δημοσιονομική πολιτική. Ο κύριος Τρισέ και εγώ και ο κύριος Σαλμούνια κάναμε ένα ταξίδι στο Πεκίνο τον Νοέμβριο του 2008 για να συζητήσουμε με τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας τα, τα, τα διάφορα προβλήματα που παραμένουν σε κρεμότητα και που θα παραμείνουν σε κρεμότητα και μετά το, την έξοδο από την κρίση και θα έχουμε έναν διάλογο με την Κίνα στα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Δεύτερη ομάδα ερωτήσεων, λέει η κυρία Περές, ο κύριος Όλι Σμιτ και μετά ο κύριος Γκαρσία Μαργάιο. Κύριος Όλι Σμιτ. Ευχαριστώ. Η ερώτησή μου κύριε Γιούνκερ αναφέρεται στις ε, χώρες εκείνες οι οποίες έχουν κειμενόμενο νόμισμα. Ασκούστηκαν κριτικές και μάλιστα και σήμερα σε εφημερίδες ότι οι Φιλανδοί επιχειρηματίες παραπονούνται για το γεγονός ότι οι Σουηδοί μπορούν να υποτιμούν το νομισμά τους κατά 5% περίπου και τα συνδικάτα στην Ευρώπη βγαίνουν και λένε ότι αυτά τα κειμενόμενα νομίσματα μπορούν να θεωρηθούν ως δημόσια, δημόσια ενισχύσεις, κρατική βοήθεια. Πώς σχολιάζετε εσείς τις κριτικές αυτές και η τρέχουσα συγκυρία σε ορισμένες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να σηκώσει ορισμένες χώρες να έχουν κειμενόμενα νομίσματα συναλλαγματικές ισοτιμίες κειμενόμενες δηλαδή και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ίσως μάλιστα και μέσα στην ομάδα ευρώ. Γκαρσία Μαργάγιο. Ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Γιούνκερς που ήρθε στην ε, συνεδρίασή μας. Έχω ένα σχόλιο πρώτα. Ένα σχόλιο πρώτα. Η διάσκεψη για την ε, απασχόληση. Κανονικά θα, γίνουν δύο διασκέψεις. Μία για τα χρηματιστήρια και μία για την ε, πραγματική οικονομία και θα γίνει και συνάντηση της Τρόικα. Ίσως επιστρέψουμε σε μια κατάσταση που ε, είχε, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από το 1996, όπου η απασχόληση ήταν καθαρά θέμα δημοδιότητας των χωρών μελών. Αλλά η ερώτηση τώρα, θεωρείτε ότι υπάρχει κίνδυνος πληθωρισμού σε οποιαδήποτε από τις χώρες της Ευρωομάδας. Δεύτερη ερώτηση. Τα τοξικά ε, προϊόντα ή ε, τοξικά περιουσιακά στοιχεία. Για τι ποσοστό μιλούμε, για πόσα μιλούμε και πώς αξιολογείται το ποσό αυτό, πώς το υπολογίζεται. Θα ε, θεωρηθεί κόστος, δηλαδή στο έτος αγοράς των ε, τοξικών αυτών περιουσιακών στοιχείων. Θα υπολογιστούν με αυτή τη βάση. Τρίτον, οι διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος για έξι κράτη-μέλη. Το Συμβούλιο θα κρίνει, θα αξιολογήσει δηλαδή την ποιότητα των δημοσιονομικών μέτρων δαπάνες ή μείωση δαπανών για την βιωσιμότητα της συνοχής και των δημοσίων της σύγκλησης και των δημοσίων οικονομικών είπατε ότι υπάρχει ζωή και μετά την, την κρίση και ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση για την περίοδο μετά από αυτή την κρίση. Θεωρείτε σκόπιμο ότι η κατανομής των πόρων συνοχής θα πρέπει να γίνεται βάση αποκριστικά του ποσοστού του ΑΕΠ ή να συμπεριλάβουμε και άλλες δύο ε, διαστάσεις της Λισαβόνας που είναι ε, το τεχνολογικό έλλειμμα και το ποσοστό ανεργίας. Αυτά και σταματώ. Ο κύριος Γκέμπελς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μας είπατε κύριε πρόεδρε του Eurogroup ότι η οικονομική κατάσταση επιδεινώνεται ολόνα και περισσότερο. Στην Ευρώπη και ότι ε, από ό,τι φαίνεται αυτό το, η αυτή η εργαλειοθήκη δεν έχει και πολλά πράγματα μέσα. Έχω την εντύπωση ότι ως επικεφαλής θα πρέπει να ακολουθήσετε την, το στρατό σας, ιδιαίτερα το γερμανικό στρατό που επιμένει να τηρηθούν οι διατάξεις του Σύμφωνου Σταθερότητας. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, το Σύμφωνο Σταθερότητας αρχίζει να λειτουργεί ως εμβαλωματική λύση. Εσείς είπατε ότι η Ευρώπη δεν πράττει αρκετά. Αυτό το περιώνυμο πλάνο ανάκαμψης των 5 δις αποφασίστηκε για δεύτερη φορά, ενώ μέχρι τώρα μόνο 3 δις ευρώ διαθέσιμων πιστώσεων έχουν βρεθεί. Τα άλλα δύο τα ψάχνουμε. Ακούμε επιπλέον κάποιους ηγέτες... ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, τον κύριο Μπράουν για παράδειγμα, που την περασμένη εβδομάδα είπε στο κοινόπιον των βουλευτών του Κοινοβουλίου οι Αμερικανοί, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και όλοι οι άλλοι έχουν δίκιο που λένε ότι δεν κάνει αρκετά η Ευρώπη και ότι όλα θα τα ρυθμίσει το G20. Μήπως έχουμε καθυστερήσει μία μάχη, μήπως δηλαδή παλεύουμε σε λάθος μάχη. Λέμε ότι η Ευρώπη έχει κάνει αρκετά στο νομισματικό τομέα, αλλά η εντύπωση που υπάρχει είναι ότι μερικές φορές δεν πιστεύετε εσείς ο ίδιος αυτά που λέτε. αγαπητέ φίλε, νομίζετε ότι με ξέρετε. Λάθος κάνετε μερικές φορές. Όταν ήσασταν μέλος της κυβέρνησης, διαπιστώνετε, έχετε διαπιστώσει ωστόσο ότι ο αρχηγός, ο επικεφαλής μιας κυβέρνησης συχνά είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί τις δυνάμεις του, αλλά αυτό συχνά οδηγεί σε κακή κατεύθυνση. Είπα εδώ και αλλού ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Eurogroup αποφάσισαν ότι δεν υπάρχει κανένας άμεσος όγκος, λόγος να αυξήσουμε τον όγκο της, του χρέους της Ευρώπης. Δεν είναι δική μου ιδέα. Όλοι το λένε αυτό και ο Gordon Brown που είπαν και επανέλαβαν αυτό. Νομίζω ότι θα ήταν λάθος να ξεκινούμε κάθε τρεις μήνες ένα καινούριο πλάνο ανάκαψης. Ας περιμένουμε τα αποτελέσματα, ας δούμε τον αντίκτυπο και μετά ας επανεξετάσουμε στα μέσα του 2010 την κατάσταση συνολικά και ας λάβουμε νέες αποφάσεις αν χρειαστούν. Δεν βλέπω γιατί πρέπει να ε, δημιουργήσουμε μια κρίση με λόγο της ε, επαναληπτικής, επαναληπτικής χρήσης προγραμμάτων ανάκαμψης. Δεν βλέπω το λόγο. Επέκρινα το μικρό μέγεθος της καθαρά ευρωπαϊκής συνεισφοράς στο πρόγραμμα ανάκαμψης. Το βέβαια, ο προπολογισμό της Ένωσης θα δώσει ο προϋπολογισμός του δίνει 5 δις. Αυτό είπα και είπα ότι είναι, είναι λίγο. Επίσης είπα ότι τα 10 15 δις από τον κοινωνικό από τον κοινωνικό προϋπολογισμό δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ε, ένας νέος κύκλος ανά, προγράμματος ανάκαμψης. Ούτως ή άλλως ο Ευρωπαϊκό προϋπολογισμός είναι περιορισμένο, Δεν έχουμε εργαλεία για να χρησιμοποιήσουμε για του τόσο τεράστιου στόχους που θέσουμε. Μετά η Ευρώπη, η ΕΠΑ, η Ιαπωνία αύξησαν τα κονδύλια, τους πόρους του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Εμείς συμβάλαμε κατά 75 δις στην αύξηση των πόρων του Ταμείου. Δεν είναι μικρή η ποσότητα. Σε ό,τι αφορά το θέμα των, των κειμενόμενων ισοτιμιών, το συζητάμε, το ξανασυζητάμε, αλλά πού είναι το, το πώς βλέπω, που, που, υπάρχει το πρόβλημα κατά την άποψή μου. Δεν πιστεύω ότι η ζώνη ευρώ θα πρέπει να επικρίνει τις χώρες της Ένωσης που διατηρούν ένα σύστημα κειμενόμενων ισοτιμιών, αλλά αποδεικνύει ότι θα ήταν πολύ πιο φρόνιμο όλα τα κράτη της Ένωσης να ήταν μέλη της ζώνης του ευρώ. Γιατί εδώ, στη ζώνη, δεν θα είχαμε τα προβλήματα που αναφέρατε. Κατόπιν, σε ό,τι αναφέρεται τα τοξικά προϊόντα, πιστεύω ότι αν δεν αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με ικανοποιητικό τρόπο, δεν θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την τα κανονική ροή των πιστώσεων. Θα υπάρχουν τα προβλήματα και οι επιφυλάξεις που προκύπτουν από το γεγονός ότι υπάρχουν ε, επισφαλής, ε, επισφαλή προϊόντα και η, ενώ η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα, ο κίνδυνος θα παραμένει. οι καθοδητήριες γραμμές που θα διευθετήσει, που θα ευθυγραμμίσει η Επιτροπή θα παρουσιαστούν αλλά δεν θα δώσουν τεχνικές λύσεις, πώς θα αποτιμώνται αυτά τα τοξικά προϊόντα, πώς ε, θα μειωθούν οι στρεβλώσεις μεταξύ τραπεζικών και μη τραπεζικών ιδρυμάτων. Υπάρχουν χώρες στη ζώνη ευρώ που έχουν ένα τραπεζικό σύστημα που περιλαμβάνει πολύ περιορισμένα τοξικά προϊόντα ενώ σε άλλες χώρες είναι κρύβονται αυτά τα προϊόντα. Θα, οι τράπεζες που έχουν καλή διαχείριση και που δεν έχουν τόσα τοξικά προϊόντα θα πληγούν ή θα ε, επενεθούν για τη συμπεριφορά τους. Δηλαδή θα, θα επιβαρύνουμε τις τράπεζες αυτές είχα προτείνει στον Επίτροπο Σπίτλα, με ρωτήσετε και για τα διάφορα διαφορετικά ταμεία, ταμείο συνοχής, κοινωνικό ταμείο, να προετοιμάσει για την Σύνοδο Κορυφή για τα κοινωνικά θέματα του Μαΐου στην Πράγα κάποιες νέες ιδέες για την κατανομή των δημοσιονομικών μέσων με των διαφόρων διαφορετικών ταμείων. Ελπίζω ο κύριος Σπίτλα που ζήτησε να με δει να κάνει αυτό που μου υποσχέθηκε ότι θα κάνει. Τι σα είπε. Κοιτάξτε, η συγκεκριμένη ερώτηση δεν είναι αν πρέπει να αγοραστούν τοξικά προϊόντα να αγοραστούν. Το θέμα είναι η σύνδεση με το σύμφωνο σταθερότητας. Που, πόσο υπολογίζονται ως δαπάνες για ποια χρονιά υπολογίζεται ως δαπάνες οι ποσότητες, την χρονιά της αγοράς ή τη χρονιά της πώλησης μείον την, ε, την απώλεια, τις ζημίες. Αυτό είναι τεχνικό ζήτημα. Άλλο τεχνικό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε πριν μπούμε σε οποιαδήποτε αντιμετώπιση των τοξικών αυτών προϊόντων. Η απάντηση δεν είναι απάντηση που μπορεί να σας δώσει ο πρόεδρος του Eurogroup. Ξέρετε ότι η Eurostat είναι αυτή που ταξινομεί τις δαπάνες. Εμείς μπορούμε να, θέσουμε, να δώσουμε μια άποψη, αλλά η Eurostat είναι αυτή που έχει την αρμοδιότητα να απαντήσει στο ερώτημά σας. Σωστό είναι το ερώτημα, γιατί οι χώρες που έχουν τράπεζες με πολλά τοξικά προϊόντα κινδυνεύουν να πέσουν θύματα υπερβολικού ελλείμματος γιατί θα απάντησαν στο ζήτημα του ότι χρειάζεται να αντιμετωπιστούν τα τοξικά προϊόντα. Αυτό όμως τόσο είναι ένα τεχνικό ζήτημα που θα πρέπει να απαντηθεί. Ευχαριστώ. Στην τρίτη ομάδα η κυρία Μαρκερίτα Στάκενβίτσα και, και μετά ο κύριος Χόπενστατ. Ε, merci, Madame la Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν πρόκειται να ρωτήσω εγώ για την Ευρωζώνη. Ε, είναι, ε, θεωρώ ότι είναι κρίμα γιατί η χώρα μου δεν μπόρεσε να μπει στην Ευρωζώνη κατά τη διάρκεια της δικής μου θητείας, αλλά ελπίζω ότι στο μέλλον θα είμαστε σε θέση να το κάνουμε. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι η Ευρωομάδα έχει έναν ηγέτη, έχει οικονομική και δημοσιονομική επιτροπή που ασχολείται με κάποια θέματα και για τις χώρες ε, που δεν ανήκουν στην, ε, Ευρωζώνη ε, η κατάσταση δεν είναι και τόσο σαφής. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και στην, εδώ στο Κοινοβούλιο ε, είμαστε υποψήφοι και για εθνικά αξιώματα, άρα αυτή τη στιγμή... Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε σε ποιον να απευθύνουμε ε, τα αιτήματά μας για να επιληθούν κάποια προβλήματα. Έχουμε ένα ταμείο για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των πληρωμών των, ε, του ισοζυγίου και θα πρέπει να υιοθετηθούν κάποια μέτρα για να αυξήσουμε τη ρευστότητα κτλ. Αυτά τα προβλήματα διακυβέρνησης αν θέλετε. Πώς θα αντιμετωπίζετε σε, οριζόντια, σε οριζόντιο επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για τα κράτη που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη. Ο κύριος Χόπενστέτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τρεις ερωτήσεις, αφού πρώτα κάνω μία παρατήρηση δεν θα επανέλθω ως υποψήφιος. 20 χρόνια Βρυξέλλες αρκούν. Όταν έρχεται ο κύριος Γιούνκερ θα προσπαθώ να έρχομαι και εγώ ως προσκεκριμένος. Ερωτήσεις. Εμπλεκόμαστε ε, σημαντικά στην ε, αναθεώρηση των hedge funds, hedge funds λοιπά Και όπως το παρελθόν με την έκθεση Λαμφαλουσί, τώρα ε, έχουμε και σωστή παροχή συμβουλών. Το ερώτημα είναι, είναι αρκετά ταχεία η αντίδρασή μας στην Ευρώπη και πώς ε, συνεργαζόμαστε με την Αμερικανική κυβέρνηση. Μήπως εμείς δεν αντιδρούμε αρκετά ταχαίως, μήπως ερχόμαστε καθυστερημένοι μετά από αυτούς. Πώς το κρίνετε αυτό. Δεύτερον, βουλώνουμε τρύπες ή σβήνουμε φωτιές. Υπάρχουν ορατές παράλληλες επαρκείς επενδύσεις σε δομές όπως οι μεταφορές, η ενέργεια. Και το τρίτο ερώτημα που εν μέρει έχει απαντηθεί, ανησυχούμε όλοι γενικά για τα όσα συμβαίνουν σε ορισμένες χώρες μέλη της Ένωσης αλλά και στην Ουκρανία. Αδυναμία πληρωμών των Ουκρανών στην οποία θα καταλήξουν πολύ σύντομα σε λίγες εβδομάδες. Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προωθεί ένα ποσό 170 εκατομμυρίων μάλλον. Ε, λαμβάνονται και άλλα μέτρα ή προετοιμάζονται και άλλα μέτρα. Και πώς συζητούνται τα θέματα αυτά μέσα στα πλαίσια της Ευρωομάδας. Βαντενμπουργκ, ευχαριστώ. Και εγώ συγκαταλέγομαι μεταξύ εκείνων που δεν θα επανέλθουν. Δέκα χρόνια αρκούν για μένα κύριε Χόπινστετ. Αλλά εκτιμώ πολύ και επιθυμώ να το εκφράσω αυτό κάθε συνεργασία που είχαμε μαζί σας στην παρούσα Επιτροπή και ιδιαίτερα για θέματα ε, της εξελίξεως ε, μισθών που ορισμένες φορές μας ε, βοηθήσατε με πολύ ευφυείς παρατηρήσεις και ίσως μπορείτε να πείτε κάτι και εν προκειμένου, δηλαδή στο πλαίσιο της παρούσας κατάστασης εξακολουθούμε να είμαστε πολιτικοί και εσείς και στην πολιτική σας οικογένεια της Ολλανδίας θεωρούμε, θεωρούν αυτοί ακόμη ότι η συγκράτηση των μισθών μπορεί να αποτελέσει το κατεξοχήν εργαλείο για την αντιμετώπιση της κρίσης. Πώς εκτιμάτε τις εξελίξεις αυτές και πώς συνδέονται με άλλα θέματα και μέσα στην προσπάθεια λήψεως μέτρων για την ανάκαμψη. Και σε ό,τι αφορά την ηγεσία της Ευρωομάδας, και τη συζήτηση που κάνατε με τον γείτονά μου κύριο Γκέμπελς εδώ. Νομίζω, ή εν πάση περιπτώσει πρέπει να οφείλουμε να σημειώσουμε ότι υπάρχει έλλειψη ηγεσία, κυρίω ό,τι αφορά τον συντονισμό των μέτρων που λαμβάνονται. Γνωρίζω ότι οι εθνικέ κυβερνήσει είναι αυτέ που ασκούν την ε, αρμοδιότητα για τον προπολογισμό. <clears throat> Αλλά πώς, έχει σημασία και αυτό, πώς γίνεται το μείγμα αυτό μέτρων που μπορούν να αποδώσουν και πώς μπορεί να συμβάλλει η Ένωση στα μέτρα που λαμβάνουν οι χώρες μέλη. Λείπει λοιπόν αυτός ο βελτιωμένος συντονισμός και ελπίζω ότι θα γίνει κάποια προσπάθεια να βελτιωθεί η κατάσταση αυτή. Μιλήσατε ήδη για τα ευρωομόλογα θεωρώ ότι αυτά συνδέονται και με το Σύμφωνο Σταθερότητας και ε, με την προσπάθεια να μειωθούν τα ελλείμματα και η χρέωση. Αυτό είναι το ένα σημαντικό στοιχείο. Το άλλο είναι η απασχόληση. Είπατε και εσείς ότι λυπήστε που δεν έγινε τέλη διάσκεψη κορυφής για την απασχόληση. Και είναι θέμα βέβαια και αυτό συντονισμού και πρόληψης ε, της τρέβλωσης του ανταγωνισμού ε, και μεταξύ χωρών οι οποίες έχουν, ε, κάνει, έχουν λάβει μέτρα, έχουν κάνει σχέδια για την αντιμετώπιση των απολύσεων. Και βέβαια οι επιχειρήσεις κοιτούν τι γίνεται στις διάφορες χώρες μέλη και σχεδιάζουν τη στρατηγική τους ανάλογα με τα μέτρα που λαμβάνονται στις διάφορες χώρες μέλη. Και αυτό πάλι οδηγεί σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Καλά, θα αρκεστώ σε αυτά τα θέματα όπου θα ήθελα να σχολιάσετε. Θα ήθελα να επανέλθω εν συντομία στην κοινωνική σύνοδο κορυφής, αυτή που σας είπα ότι λυπήθηκα γιατί μίκρινε αν θέλετε η σύνθεση. Ε, ήθελα να σας πω ότι και εγώ ανησυχούσα και για τα αποτελέσματα ε, μιας τέτοιας κοινωνικής ε, συνόδου. Ε, εάν συνεδριάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 27 κράτη-μέλη στην Πράγα για να συζητήσουν τα θέματα αυτά χωρίς απτό αποτέλεσμα, χωρίς συγκεκριμένο αποτέλεσμα, η κατάσταση θα ήταν φρικτή θα έλεγα. Δηλαδή θα πρέπει τα κράτη-μέλη, οι κυβερνήσεις να κάνουν μια λεπτομερή προετοιμασία εκ των προτέρων και μετά να γίνει η σύνοδος αυτή κορυφής. Πραγματικά αν δεν γινόταν κάτι τέτοιο θα ήταν ε, πραγματικά κρίμα. Όμως από τη στιγμή που έγινε αυτή η πρόσκληση και για να γίνει αυτή η σύνοδος, όντως θεωρώ ότι το, το μήνυμα που στείλαμε ακυρώνοντάς το ή υιοθετώντα μια νέα διάσταση τέλο πάντων είναι ε, λυπηρό. Και το είχα συζητήσει και με τον Επίτροπο τον κύριο Σπίτλα. Ε, είχαμε πει ότι θα πρέπει να, οι κατευθυντήριες γραμμές που υιοθετήσαμε το 1997 θα πρέπει να επανεξεταστούν και να, και να αλλάξουν, να προσαρμοστούν. Και ελπίζω να το κάνει αυτό η Τρόικα, διότι δεν θα είμαστε και 27 εκεί, αλλά τέλος πάντων κάτι χρειάζεται να γίνει. Τώρα, όσον αφορά το συντονισμό, που είναι, αν θέλετε, και ο βασικός στόχος της, Ευρωζώ, της Ευρωομάδας. Είναι όλο ένα και πιο δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο, διότι η θέση αφετηρίες όλων των κρατών διαφέρουν. Γιατί Υπάρχουν κάποια κράτη που έχουν ε, κάπως προχωρήσει. Ε, υπάρχει μια μικρή ανάπτυξη. Ούτως ή όλως ε, η Ευρωζώνη βρίσκεται σε ύφεση αυτή τη στιγμή. Αλλά κάτι κράτη-μέλη τα οποία έχουν περιθώρια ε, ελιγμόνο στο δημοσιονομικό επίπεδο που είναι επαρκή και αρκετά. Άλλα κράτη-μέλη όμως, τα οποία ήταν, ε, συμπεριφέρθηκαν πολύ σωστά ε, στο παρελθόν, ίσως να μην έχουν τα ίδια περιθώρια. Γι' αυτό προσπαθήσαμε να υιοθετήσουμε ένα γενικότερο πλαίσιο, το κάναμε στο, στην Ευρωομάδα, το κάναμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και είπαμε ότι θα πρέπει να τονίσουμε τα θέματα των δημοσίων επενδύσεων και από εκεί και πέρα θα πρέπει τα κράτη-μέλη να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα περιορίσουν με ένα εστιασμένο τρόπο τα, ε, τις τα φορολογή, ε, τις, δημοσιονομικές τους, τα δημοσιονομικά του μέτρα. Τώρα βέβαια δεν μπορεί να είναι τα μέτρα τα ίδια, διότι οι καταστάσεις των κρατών μελών είναι διαφορετικέ Στο εσωτερικό τη ζώνη θα έχουμε ε, κράτη που θα ε, έχουν ένα έλλειμμα που θα ξεπεράσει το 17-18%. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε από την Ιρλανδία να έχει ένα πρόγραμμα ανάκαμψης ε, με άλλες χώρες που έχουν διαφορετική δημοσιονομική κατάσταση. Δεν λέω ότι είναι ευσεβή πόθο αυτό, αλλά δεν γίνεται, δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε την, τα ίδια μέτρα για όλες τις χώρες. Ο συντονισμός δεν είναι να επιβάλλουμε μία ομοιομορφία των μέτρων. Υπάρχουν διαφορετικά προγράμματα ανάκαμψης και εκεί όμως υπάρχουν αντιφάσεις, εμφανείς αντιφάσεις. Δεν υπάρχει καμία χώρα που ε, στο πρόγραμμα ανάκαμψης θα μπορούσε να, να υιοθετήσει μέτρα τα οποία θα ζημίωναν άλλες χώρες ε, ε, της ζώνης ευρώ. Επομένως, ναι, δεν υπάρχει ομοιομορφία, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν κάποια προβλήματα στα προγράμματα για το συντονισμό των προγραμμάτων ε, ανάκαμψης. Τώρα, ήθελα να πω στην, στον Φιλανδό συνάδελφο ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εγώ θεωρώ ότι είναι ζωτική σημασία να υπάρχει μια αλληλεγγύη με τις χώρες Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης την, στην, στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής αυξήσαμε την δυνατότητα και την διευκόλυνση που υπάρχει για να για το ισοζύγιο πληρωμών και η διαφορά να είναι στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και είπαμε ότι αυτό θα το κάνουμε για την ημέρα που χρειάζεται να προσφύγουμε σε ένα τέτοιο ταμείο, σε, μια σε ένα τέτοιο εργαλείο. Το κάναμε για την Ουγγαρία, για τη Λετωνία, το κάνουμε αυτή τη στιγμή για τη Ρουμανία. Είναι προφανές ότι δεν έχουμε κανένα συμφέρον εμείς αμέλη της ζώνης ευρώ να ε, εισάγουμε σοβαρούς σταθεροποιητές στο... ή αποσταθεροποιητές στην ευρωπαϊκή ζώνη. Είναι σοβαρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ε, οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και σαν σοβαρά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Τώρα, είναι διαφορετική κατάσταση για την Ευρωζώνη. Για μια χώρα που δεν είναι μέλος της ζώνης ευρώ, μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα και να δράσουμε ταχύτερα, παρότι μέσα στην ε, Ευρωζώνη. Υπάρχει ο κανόνας opt-out όμω. και αυτό δεν επιτρέπει μεγάλο περιθώριο ερμηνεών. Ε, ε, επιμένω λοιπόν στην δήλωσή μου το γεγονός ότι ε, μια χώρα της μέλο μέλος της ζώνης ευρώ ενδεχομένως θα έπαβε τι πληρωμές δεν μπορεί να γίνει, δεν θα γίνει. Αν ωστόσο γίνει πολύ σύντομα θα ήμασταν σε θέση να προσφέρουμε μια ικανοποιητική λύση. Δεν έχει νόημα να συζητούμε περισσότερο από τα ήδη λεχθέντα για τα θέματα αυτά σε δημόσιες ε, συζητήσεις γιατί πρόκειται για πάρα πολύ ε, εκρηκτικό υλικό και δεν μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει τη φωτιά με φωτιά σε ό,τι αφορά την έκθεση της ομάδας De και το εάν είναι ε, έκθεση για τις 27 χώρες μέλη και όχι για τις, ε, μόνο για τις χώρες της όλης Ευρώπης. εγώ θεωρώ ότι είναι ρεαλιστική η έκθεση και πρέπει να εφαρμοστεί αμέσως. Συμφωνώ με την ανησυχία σας ότι κινδυνεύουμε να χαθούμε σε λεπτομέρειες εάν δεν εφαρμόσουμε ταχύτατα τα όσα ήδη μπορούν να εφαρμοστούν και όπως και οι Αμερικανοί άλλωστε. Εγώ συζητώ συχνά με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών για παρόμοια θέματα και θεωρώ ότι πρέπει να εφαρμοστούν όλα τα στοιχεία που διαλαμβάνει η έκθεση Τελαρόζιε. Πρέπει να εφαρμοστούν μέχρι τέλος του έτους. Εδώ χρειάζεται πραγματικά ταχεία ε, λήψη δράσεως. Ευχαριστώ. Ο Λάζλο Μπούτσεκ και κατόπιν ο κύριος Ροζάτη. Ευχαριστώ πρόεδρε μία παρατήρηση για την ανθεκτικότητα. Εγώ προέρχομαι από μία, από μία χώρα εκτός της ζώνης ευρώ. Σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις που θα λόγω του ότι δεν μπορούμε να ε, μπούμε στη ζώνη ευρώ, ευρώ εφόσον δεν πληρούμε τα κριτήρια του Μάστερ, συμφωνώ μαζί σου. Αλλά σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, τι θα κάνετε θα κάνετε το ίδιο και στα κράτη που είναι στη ζώνη ευρώ αλλά δεν πληρώνουν τα κριτήρια. Αυτό θα ήθελα να το ζητήσω για να το δω για να δείτε μια συνέπεια στις θέσεις σας. Για τα κράτη εκτός ζώνης ευρώ. Θα ήθελα να πω το εξή. Στην περιοχή μας, στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, το κύριο πρόβλημα και τροτότητας ήταν το τεράστιο ισοζύγιο των χρυσών συναλλαγών και ένα, μία από τις αιτίε ήταν η ελεύθερη ροή κεφαλαίων. Ο τεράστιος επαναπατρισμός κεφαλαίων που έφυγαν για άλλη χώρα τα τελευταία δύο-τρία χρόνια. Σε εμά μιλάμε για 8 δις. Επιπλέον υπάρχει μια υποτίμηση του νομίσματος. Δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τα φορολογικά κίνητα γιατί ήμασταν πιο ευάλωτοι από άλλους. Θέλουμε να μπούμε στην Ευρωζώνη. Το ερώτημα είναι πώς μπορούν να μας βοηθήσουν τα κράτη της Ευρωζώνης. Μπορούν να σταματήσουν μια κατάσταση στην οποία μας παραπέμπουν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όπως σαν ήμασταν το Πακιστάν. Ξέρουμε το θέμα των 15 δις, αλλά στα πλαίσια της αλληλεγγύης που αναφέρεται, θα έπρεπε η πρακτική παραπομπή στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο να πάψει. Δεύτερον, μπορεί να βοηθήσει με μέτρα ρευστότητα η Ευρωζώνη. Η, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χορηγεί ρευστότητα μόνο στην Ευρωζώνη. Αυτό είναι διακριτική μεταχείριση. Πώς μπορεί να μας βοηθήσει ε, η Ευρωζώνη να μπούμε στο, ε, στο, στο δεύτερο μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών, αν μη τι άλλο. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε. Μπορείτε να μας βοηθήσετε τουλάχιστον ή πρέπει μόνοι μας να τα κάνουμε όλα. Ευχαριστώ. Merci, Darius Rosati, puis Astrid Luling. Darius Rosati και μετά Astrid Luling. Ευχαριστώ. Για το θέμα του μεγέθους του, των φορολογικών κινήτων. Ξέρω ότι η Ευρώπη είναι σε διαφορετική κατάσταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μην ξεχνάτε ότι αυτό θα πρέπει να, τα φορολογικά κίνητα πρέπει να αντισταθμίζουν τη μείωση της ζήτησης. Θεωρείτε ότι από αυτή την άποψη τα κίνητρα είναι παρκή. Όχι για το αν υπάρξουν η αύξηση του χρέους με αρνητικές μελλοντικές συνέπειες. Θεωρείτε ότι κάνουμε αρκετά σε ό,τι αφορά τα φορολογικά κίνητρα για να ε, αντισταθμίσουμε την μείωση της ιδιωτική ζήτησης. Διαφωνώ επίσης μαζί σας όταν είπατε ότι το πιο σημαντικό θέμα που υποκρύπτεται στην ύφεση στην Ευρώπη είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης και ότι η άμεση προτεραιότητα θα ήταν η αποκατάσταση αυτή της εμπιστοσύνης. Το ερώτημα προς εσάς είναι το εξής. Πώς ερμηνεύετε τις αιτίες και τους λόγους της κατάρρευσης του πιστοτικού της πιστοτικής κατάρρευσης στην Ευρώπη. Μήπως αυτό, αυτό οφείλεται στην έλλειψη ρευστότητας. Αν ναι, μήπως έπρεπε να είναι πιο δραστήρια η κεντρική τράπεζα. Αν αρκεί η ρευστότητα, και εγώ πιστεύω ότι αρκεί στο σύστημα τώρα, μήπως το πρόβλημα είναι οι τράπεζες που δεν θέλουν να ε, δανείσουν. Σε μια τέτοια περίπτωση η εμπιστοσύνη, η έλλειψη εμπιστοσύνη δηλαδή αντικατοπτρίζει ψηλό πιστοτικό κίνδυνο. Εδώ τι θα κάνουμε. Τρίτον, η έλλειψη ε, εμπιστοσύνη μπορεί να οφείλεται σε χαμηλέ μακροοικονομικέ προσδοκίε. Και εδώ οι κυβερνήσει είναι αυτέ που πρέπει να λάβουν μέτρα για να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη στο μέλλον. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα πρέπει να δαπανούμε μόνο. Θα πρέπει να, προσ... να προσβλέπουμε σε διαφορετικές μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την ε, αύξηση του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη και θα αποκαταστήσουμε έτσι την εμπιστοσύνη. Δεύτερον, τα κριτήρια του Μάστριχτ. Προέρχομαι και εγώ από ένα νέο κράτος μέλος. Θυμάμαι όταν στο Κοινοβούλιο στείλαμε ε, μία επιστολή στην καγκελάριο Μέρκελ κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Προεδρίας πριν από δύο χρόνια και ζητούσαμε να αναθεωρηθούν τα κριτήρια του Μάστριχτ. Σε εποχές παχαίων αγελάδων η απάντηση ήταν δεν έχει νόημα, δεν υπάρχει λόγο, μην πειράζουμε τα κριτήρια. Τώρα μα λέτε μην πειράζετε τα κριτήρια γιατί ο κερί είναι χαλεπή. Φοβάμαι ότι δεν θα υπάρχει ποτέ κάποια καλή στιγμή να εξετάσουμε τα κριτήρια αυτά. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι τα κριτήρια συναλλαγματική ισοτιμία που έγινε, συναλλαγματική έγινε πριν από 20 χρόνια με τελείω διαφορετικέ ε, διεθνείς συνθήκες, ούτε παγκοσμιοποίηση των οικονομικών αγορών, είτε ούτε οικονομική σταθερότητα. Μήπως μπορούμε να ξαναδούμε το ζήτημα αυτό, ίσως όχι αύριο ή μεθαύριο, αλλά να ξαναδούμε το ότι τα κριτήρια αυτά κατακρίνονται από σοβαρούς οικονομολόγους. Η κυρία Λούλινγκ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. η συνάδελφος συντονίστρια των σοσιαλιστών σας ανήγγειλε ότι αποφασίσαμε σήμερα το πρωί να πάυσουμε το σύστημα του τραπεζικού απορρίτου το 2014. Ε, σχετικό, σχετική είναι η αναγγελία αυτή. Στο μέτρο που ούτε η Επιτροπή μας, ούτε το Κοινοβούλιο είναι αυτοί που θα αποφασίσουν αυτή την αποφασία, αλλά όντω με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίναμε μία έκθεση της Επιτροπής που, θα, που ζητά το 2014 να πάυσει η παρακράτηση στην πηγή στο πλαίσιο της οδηγίας για την φορολόγηση των τόκων. τόκων. Μόνο το σύστημα ενημέρωσης θα πρέπει να υπάρχει μετά το 2014. Παρότι είναι και γραφειοκρατικό και αναποτελεσματικό. Αλλά εν τη σοφία τη, η πλειοψηφία τη Επιτροπή αποφάσισε σήμερα ότι θα έπρεπε να λάβουμε σήμερα την απόφαση αυτή να πάψει το 2014 το σύστημα που λειτουργεί καλύτερο, που είναι λιγότερο δαπανηρό και πιο αποτελεσματικό. Όταν το 2011 και ότι το 2011 θα ζητήσουμε από την Επιτροπή ούτω ή να υποβάλει μια έκθεση για να διερευνήσει πώς το σύστημα ανταλλαγών πληροφοριών θα μπορούσε να λειτουργήσει. Κάτι που δεν συμβαίνει τώρα. Επιπλέον, ε, κατά κάποιο τρόπο προτέχουμε τώρα, αλλά ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία αντίφαση του Κοινοβουλίου είναι αυτή. Θέλω απλά να διευκρινίσω τις πληροφορίες. Τώρα, στην παρουσίαση που κάνετε κύριε Πρόεδρε αναφερθήκατε στους φόβους που στους φόβους ότι μπορεί να παραμείνουν οι τεράστιες δαπάνες που έχουν ξεκινήσει τα κράτη-μέλη για τα σχέδια ανάκαμψης, δεν θα έχουν άμεσα αποτελέσματα. Στο πλαίσιο αυτό θέλω να ξέρω το εξή: Όταν αναλύεται αυτά τα σχέδια ανάκαμψης και εξετάζεται τα διάφορα κράτη της ζώνης ευρώ με βάση το κριτήριο του δημόσιου ελλείμματος διακρίνεται μεταξύ επενδυτικών δαπανών και καταναλωτικών δαπανών. Θεωρείται ότι τα κράτη οφείλουν να μεριμνούν ούτως ώστε οι καταναλωτικές δαπάνες τους να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα στα πλαίσια του προγράμματος, των προγράμματων ανάκαμψης τι συνέπειες θα έχουν οι εξελίξεις αυτές στα ελλείμματα. Σε κάποιες χώρες τα ελλείμματα φτάνουν κοντά το 10%. Ο κ. Σκουτ Λάουκ. Äh, δύο σύντομες ερωτήσεις κύριε Γιούνκερ. Πρώτη. Ρόροφ και Ράινερτ εξέτασαν 200 χρόνια τραπεζικών κρίσεων και δημοσίευσαν πρόσφατα το τι βρήκαν. Όταν μια κρίση προκύπτει από τις τράπεζες, κρατάει περισσότερο, τα διπλάσια, 3 μέχρι 6 χρόνια. Και η χρέωση, το χρέος μιας χώρας ξεκινάει από 100 πριν την κρίση και φτάνει στα 186. Οι αντιδράσεις είναι bailout και λιγότερες, λιγότερα έσοδα. Βλέπετε να διαφέρει η παρούσα κρίση από τις κρίσεις από τις τελευταίες 200. Δεύτερη ερώτηση, κατά τη γνώμη σας, πώς θα πρέπει να είναι η αρχιτεκτονική της εποπτείας και η δημοσιονομική, δηλαδή σε ό,τι αφορά την εποπτεία των τραπεζών των ασφαλιστικών εταιριών. Πρέπει να κάνουμε και κάποια εναρμόνιση στην Ευρώπη. Λέτε από τη μια μεριά ότι, χαίρε, ότι σας ικανοποιεί η Δελαροζιέρα, από την άλλη μεριά θέλετε να μείνουν οι εποπτικές αρχές σε όλες τις χώρες μέλη. Το βρίσκεται σωστό αυτό για μετά την κρίση. Πώς φαντάζεστε την αρχιτεκτονική της εποπτείας της οικονομίας μετά την κρίση. Τρεις μικρές ερωτήσεις. Πότε θεωρείτε ότι η ανάκαμψη θα εμφανιστεί, γιατί βλέπουμε κάποιες ημερομηνίε οι οποίες εξαγγέλλονται. Συμφωνείτε με τις ημερομηνίες. ποια είναι τα δικά σας προγνωστικά. Δεν λέω ότι έχετε μια ε, ε, γυάλινη μπάλα μπροστά σας, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, αυτές Εσείς πώς κρίνετε αυτές τις υψηλές αμοιβέ ε, των ε, διαφόρων διευθυνών, των, των ταμπόνους που παίρνουν οι διευθύνοντες στις μεγάλες εταιρείες. Ε, πώς κρίνετε την κατάσταση, πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να απαγορεύσει τα stock options, γιατί διάφορα κράτη-μέλη θεωρούν ότι α, τη μεγάλη τη και τα θα εγκαταλείψουν τη χώρα και θα πάνε στη διπλανή χώρα που δεν εφαρμόζει τέτοιου είδους ε, μέτρα. Τώρα, Τελευταία ερώτηση για τα ευρωομόλογα. Είναι μεγάλη συζήτηση, ε, υπάρχουν πολλές πτυχές. Ε, ο Ντελόρ είχε πει ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ήταν καλό γιατί θα υπήρχε ανάκαμψη των δημοσίων επενδύσεων και εάν υιοθετήσουμε αυτά τα ευρωομόλογα, δημιουργήσουμε αυτά τα ευρωομόλογα για να περιορίσουμε το spread στο, στο ιστορικό της ζώνης ε, ευρώ, θα πρέπει να υπάρξουν, να αποφασίσουμε και τα κριτήρια για την χορήγηση τέτοιων ή τέτοιου είδους διευκολύνσεων ε, πληρωμών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα ή η Ευρωομάδα έχει την αρμοδιότητα να διαχειριστεί αυτά τα ευρωομόλογα και αν όχι, τι ε, πρωτοβούλια πρέπει να αναλυφθεί για να υπάρξει αυτή η αρμοδιότητα. Α πούμε, παραδείγματο χάρη όταν το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο δανείζει χρήματα, ε, υιοθετεί κάποιε ε, προδιαγραφέ, κάποιε προποθέσει. Εμεί δεν τι έχουμε αυτέ τι προποθέσει. Αν θέλουμε να το κάνουμε, πώ θα ξεκινήσει αυτή η πρωτοβουλία. Θα ξεκινήσω, κυρία Πρόεδρε, με τις δικές σας ερωτήσεις για τα ευρωομόλογα. Σας είπα αυτά τα οποία εγώ πιστεύω. Διότι θεωρώ, διαπιστώνω, ότι ο ενθουσιασμός των κυβερνήσεων για να εφαρμόσουν τέτοιου είδους, ένα τέτοιο είδους μηχανισμό, μια τέτοιου είδους διευκόλυνση. Ο ενθουσιασμός δεν ξεχυλίζει και δεν μπορώ να καταλάβω τι πρωτοβουλία θα μπορούσαμε να ζητήσουμε εμείς στην Ευρωομάδα, στο Eurogroup, διότι υπάρχουν τρεις φανατικοί οι οποίοι στρέφουν τα πειρά τους εναντίον μου κάθε φορά που ανοίγω το στόμα και λέω κάτι υπέρ των ευρωομολόγων και κάποια από αυτές είναι μια κυρία, μια κυρία ε, από τη χώρα σας που δεν ε, ανήκει στη δική μου ε, πολιτική ομάδα. Τέλος πάντων, εγώ θα συνεχίσω ε, να επιμένω στην ιδέα μου, θα το συζητώ και στην Επιτροπή και στην Κεντρική Τράπεζα, διότι πιστεύω ότι θα έρθει η μέρα που θα έχουμε ένα τέτοιο εργαλείο στη διάθεσή μας, διότι πραγματικά θα το έχουμε ανάγκη. Και μεγάλη ανάγκη κιόλας. Τώρα, το σύστημα των αμοιβών των σου αυτά που πρέπει να επανεξεταστούν, αυτά γίνον, θα πρέπει να γίνουν σε εθνικό επίπεδο. Δεν μπορώ να φανταστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντάσει ή να προτείνει μια οδηγία για το θέμα αυτό. Δεν υπάρχει, μπορεί να υπάρχει σκοπιμότητα να ε, υιοθετήσει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές η Κομισιόν για να πλησιώσει μια ζήτηση που θα γίνει σε εθνικό επίπεδο. Και όταν πριν από τέσσερα χρόνια ξεκίνησε αυτή τη συζήτηση, κανείς δεν ήθελε να το ακούσει. Ενώ τώρα όλοι διαρριχνύουν τα ημάτια τους και θέλουν να υιοθετήσουν τέτοιου είδου συστήματα επανεξέτασης αυτών των υπερβολικών αμοιβών. Τώρα, η ανάκαμψη θα είναι πολύ μικρή, πολύ μικρή και θα παραπέει το 2010. Από το 2011 όμως θα γίνει κάποια, θα γίνει κατάσταση θα εμφανιστεί πιο στιβαρή αν θέλετε, αλλά για αρκετά χρόνια ακόμα θα ασχολούμεθα με τις συνέπειες της κρίσης. Τώρα, άλλες ερωτήσεις. Θα πρέπει να δώσω μία σύντομη απάντηση, διότι θα πρέπει σε δύο λεπτά να φύγω. Η κυρία Λούλινγκ έδωσε κάποιες χρήσιμες διευκρινήσεις για το τραπεζικό απόρριτο και για τις ανταλλαγές πληροφοριών. Τον την ευχαριστώ. Απλώς ήθελα να πω ότι όταν θα, όταν θα εξετάσουμε τις περιπτώσεις των χωρών που θα αποκλίνουν από τα υπερβολικά ελλείμματα, στο, κριτήριο των υπερβολικών ε, ελλημάτων, εξετάζουμε ε, ξεχωριστά τις διάφορες δαπάνες, αλλά και το πώς, πώς ε, λειτουργούν και τι συνέπεια έχουν οι αυτόματοι σταθεροποιητές. Διότι πρέπει να δούμε το έλλειμμα οφείλεται στην ε, εφαρμογή, στην αυτόματη εφαρμογή των σταθεροποιητών ή οφείλεται σε, άλλους, σε άλλες δαπάνες. Τώρα, κύριε Ροζάτη, δεν μπορούμε να επανέλθουμε στα κριτήρια σύγκλησης. Έχετε κάνει, έχετε κάνει πολλά έργα, έχετε αφιερώσει πολλά έργα για την Οικονομική Ένωση και Νομισματική Ένωση. Δεν μπορούμε τώρα όσα έχουμε κάνει στο παρελθόν να τα αναθεωρήσουμε, να τα ανασκευάσουμε και να αλλάξουμε τα κριτήρια. Διότι υπάρχει συνθήκη, τελείωσε τώρα αυτό η, παρατή, συμμόρφωση, αν θέλετε, με, την, με τα κριτήρια αυτά σύγκλησης και τα κριτήρια προσχώρησης στην Ευρωζώνη επέτρεψαν να φτάσουμε σε ένα επίπεδο σταθερότητας και ορίμανσης που μας επέτρεψε να διατηρήσουμε την αξιοπιστία μας στις διεθνείς αγορές. Δεν μπορούμε επομένως να επανέλθουμε και να αλλάξουμε αυτά τα κριτήρια και παραδέχομαι βέβαια ότι κάποια αυτά τα κριτήρια χρειάζεται να επανεξεταστούν. Όμως επί του παρόντος δεν μπορούμε να το κάνουμε. Επίσης ήθελα να πω στους φίλους μας ε, της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης ε, ότι δεν ε, θεωρώ ότι δημιουργούν ένα μπλοκ, ότι αποτελούν ένα μπλοκ. Ήδη εμείς έχουμε διαθετήσει κάποια μέτρα για να βοηθήσουμε τις χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα σαν και αυτά τα οποία αναφέρεται. Αυξήσαμε την διευκόλυνση των 25 από 25 σε 50 δισεκατομμύρια ε, και είπαμε ότι είμαστε διατεθειμένοι και κατά τα λοιπά ε, να επιτρέψουμε μία προσέγγιση με τη ζώνη ευρώ και θα πρέπει από καιρό σε καιρό στην Ευρωομάδα να προσκαλούμε κάποιες χώρες που δεν ανήκουν στη ζώνη ευρώ για να μπορέσουμε να συγκλίνουμε τις, ε, τις θέσεις μας. Ε, δεν θέλω, δεν μπορώ, δυστυχώς δεν μπορώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις γιατί πρέπει να φύγω. Να, προσθέσω, να προσθέσω μόνο κύριε Λάουκ ότι συμφωνώ με τις βασικές γραμμές της εκθέσεως Λαροζιέρ. Συμφωνώ και ε, με την ιδέα να παραμείνουν οι 27 εποπτικές αρχές, ε, γιατί προκλήθηκε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τις τράπεζες, για τις ε, μητρικές τράπεζες και τις θηγατρικές σε άλλες χώρες. Γι' αυτό και θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν 27 εποπτικές αρχές. Όμως αυτές οι 27 εποπτικές αρχές θα πρέπει να ακολουθούν ενίους κανόνες. Σας ευχαριστούμε πραγματικά κύριε Πρόεδρε για την πιστή παρουσία σας εδώ. Δεν ξέρω πώς θα είναι το επόμενο κοινοβούλιο, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να συζητήσουμε αυτή την τόσο καλοποφόρα συνεργασία μας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Μισό λεπτό κύριοι συνάδελφοι, μην φύγετε. Όπως ε, είχαμε συμφωνήσει μετά από αίτημα της κυρίας Στακεβιτσιούτερ, όσοι θέλουν θα βγάλουμε μια φωτογραφία. Ελάτε λοιπόν όλοι κάτω για να βγούμε μια αναμνηστική φωτογραφία.